Hello everyone. Καλημέρα σας και πάλι. Ξεκινούμε την απογευματινή μας συζήτηση. Είναι χαρά μου να καλωσορίσω την Υπουργό Μπέατε Χάρτιγκερ Κλάιν, Υπουργό Εργασία, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών τη Αυστρία στη συνεδρίασή μα σήμερα. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Αυστρία για την ανάληψη της τρίτης Προεδρίας του Συμβουλίου μετά την επιτυχή Προεδρία τους το 1998 και το 2006. Το μότο της ε, Προεδρίας είναι «Η Ευρώπη που προστατεύει» και βεβαίως είναι μια έμπνευση για όλους μας. Οπότε υπό το φως αυτό θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία για το επόμενο εξάμεινο στην ε, Προεδρία σας. Η Προεδρία η Αυστρία αναλαμβάνει την Προεδρία λίγο πριν τι ε, ευρωεκλογέ και πραγματικά είναι μεγάλη πρόκληση για να κλείσουν πολύ σημαντικοί φάκελοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεργαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο μαζί σα ώστε αυτό να καταστεί δυνατό. Ήδη έχουμε κάποιε ενδείξει. Οπότε Κυρία Υπουργέ, θα μιλήσετε για πράγματα όχι μόνο του δικού σας χαρτοφυλακίου, αλλά και για το κλίμα και για, την, ε, ε, για το περιβάλλον, γιατί ο, η Υπουργό και δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Ε, ως συνήθως λοιπόν, αρχικά η υπουργό θα καθορίσει τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας και μετά θα κάνουμε μία συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας για διάφορα σημεία κλειδιά. Πριν δώσω το λόγο στην Υπουργό, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερω εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, το θέμα της, ε, του προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να συμπεριληφθεί το πρόγραμμα για την υγεία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus. Και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος, διότι οι στόχοι των ταμείων και των προγραμμάτων ε, της, ε, των κοινωνικών τομέων και της εργασίας είναι τελείως διαφορετική από αυτούς της υγείας και στο παρελθόν με πολύ περιορισμένους ε, πόρους είχαμε επιφέρει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της Ευρώπης και θεωρούμε ότι ένα τέτοιο μικρό πρόγραμμα όπως είναι το πρόγραμμα για την υγεία θα χαθεί μέσα στο, θα χάσει την ορατότητά του, την επιρροή του αν ενταχθεί σε ένα μεγάλο ταμείο 20 φορέ μεγαλύτερο από το ίδιο. Οπότε θα θέλαμε να βγει το πρόγραμμα υγείας από το κοινωνικό ταμείο Plus και να παραμείνει ξεχωριστό και ζητούμε βεβαίως την ε, στήριξη και της προεδρία αλλά και των κρατών μελών για το σημαντικό αυτό θέμα. Οπότε, χωρίς να μιλήσω εγώ άλλο, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, ε, αγαπητοί συντονιστές, αγαπητά μέλη της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί δερμηνείς, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, παρουσιάσω σήμερα τις ε, προτεραιότητες της, Ευρωπαϊκής, της Αυστριακής Προεδρίας για τον τομέα της υγείας, φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα, την ασφάλεια τροφίμων, την, τα θέματα του κλίματος και του περιβάλλοντος. Αυτό το ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα θεμάτων προκύπτει διότι ε, εγώ εκτός από τα δικά μου θέματα, του δικού μου χαρτοφυλακίου, θα σας παρουσιάσω και τα χαρτοφυλάκια δύο ακόμα υπουργών, της ε, Υπουργού Κιώστιγκερ, Ελίζαμπεθ η οποία είναι υπεύθυνη για, το, για τα θέματα κλίματος και περιβάλλοντος, η οποία στις 8 ε, Ιουλίου μπορώ να σας ανακοινώσω ότι γέννησε το γιο της, οπότε βρίσκεται σε άδεια μητρότητας. Οπότε θα παρουσιάσω εγώ τα δικά της θέματα και βεβαίως ε, χαίρομαι πολύ που μπορώ να το κάνω αυτό. Επίσης θα παρουσιάσω τα ε, θέματα του Υπουργού Ιώζεφ Μόζερ που είναι υπεύθυνο για την οδηγία για την πρόθεση των ε, καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων. Για μας ως Προεδρία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νομοθέτη. Και ως προς αυτό θεωρώ ότι βεβαίω η, παρουσίασή μου θα, δοθεί, θα είναι στη διάθεσή σα για περαιτέρω μελέτη. Ακριβώ λοιπόν επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα που θέλω να σα παρουσιάσω, παρακαλώ την κατανόησή σα για το ότι μπορώ, μπορεί να μην μπορώ να σα απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα, αλλά βεβαίω θα απαντήσουμε αργότερο γραπτό. Πριν σα παρουσιάσω λοιπόν τα, τις βασικές πρωτο, προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τη δουλειά και για την υποστήριξη την Βουλγαρική Προεδρία κατά τη διάρκεια του τρίου του ε, του τρίου των Προεδριών. Η Αυστρία στις αρχές ε, Ιουλίου ανέλαβε για τρίτη φορά, όπως είπε και η Πρόεδρος, την Προεδρία του Συμβουλίου για σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Ακριβώ πριν από τι εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάιο του 2019, η γενική θέση είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερου φακέλους και αν γίνεται να του ολοκληρώσουμε. Ω συνομοθέτης, η θέση και η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, δημιουργία του Ευρωπαϊκή Πολιτική για την υγεία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον είναι φυσικά ε, θεμελιώδης σημασία. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει λοιπόν να δουλέψουν ε, συστηματικά περισσότερο από, ποτέ και ε, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για να μπορέσουν να επικεντρωθούν στις βασικές, στους βασικούς νομοθετικούς φακέλους για να βρουν από κοινού λύσεις. Βεβαίω δεν τίθεται ε, θέμα ότι η Προεδρία του Συμβουλίου μπορεί να επιτύχει η πρόοδο μόνο αν μπορέσει να βασιστεί στην ενότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών. Με την ε, Προεδρία λοιπόν του Συμβουλίου η Αυστρία προσπαθεί ω ε, ως χώρα στο κέντρο της Ευρώπη να παίξει το ρόλο του γεφυροποιού για αυτή την εξέβρεση τη Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αυστρία αναλαμβάνει βεβαίως την Προεδρία με το ε, μότο που ανέφερε και ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ στην ε, ομιλία του για την ε, κατάσταση της Ένωσης. Η Ευρώπη που προστατεύει. Στόχος είναι να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου τώρα να μπω λίγο στα τομεακά επιμέρους θέματα της Προεδρίας μας. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας θα είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η συμπερίληψη της ψηφιοποίησης. Το θέμα αυτό θα το δούμε, θα το συζητήσουμε στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Υγείας στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος στη Βιέννη. Ουσιαστικά σημεία αποτελούν ε, οι ε, φιλοδοξίες της ε, προεδρίας, της, του τρίου των προεδριών της Εστονίας, για τα, με, το, αποτελε, με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Υγεία στην ψηφιακή κοινωνία, καθώς επίσης και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενισχυμένη ψηφιακή αναδόμηση της υγείας, του τομέα της υγείας. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι το θέμα επενδύσεις στην ε, ψηφιακή, σε ένα ψηφιακό τομέα της υγείας και η χρήση δημοσίων κονδυλίων στον τομέα της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο, ο δεύτερο βασικός πυλώνας του άτυπου ε, Συμβουλίου Υπουργών θα, αποτελέσει ε, θα αποτελέσουν οι ρυθμιστικές ε, και πολιτικές προκλήσει για την ευρωπαϊκή έγκριση φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει μια συζήτηση μεταξύ των Υπουργών Υγείας και με τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής, Επιτρο... Ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων, Γκουίντο Ράζη. Στο νομοθετικό τώρα κομμάτι θα επικεντρωθούμε στους εξής φακέλους. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για, τον, για το σχέδιο κανονισμού για την αξιολόγηση των ε, τεχνολογιών υγείας που βεβαίως είμαστε ιδιαίτερος ε, θετικοί απέναντί τους και θα τα συζητήσουμε στο Συμβούλιο εντατικά. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μία ε, ενδιάμεση συνολική προσέγγιση. Ε, μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει, έχουν σχεδιαστεί μάλλον 8 συνεδριάσεις ε, ομάδων εργασίας. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα που προκύπτουν στα κρατη και θα προσπαθήσουμε με τη, επί βάση αυτή να βρούμε, με το νέο, με το, να βρούμε ένα νέο κείμενο από τα κρατη για να καλύψουμε τις ανησυχίες αυτές. Ε, γι' αυτό έχουμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ε, στείλει την, ε, μια πρόσκληση στα κρατημέλη για να μας στείλουν συγκεκριμένες προτάσεις και για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τη φιλοδοξία που έχει δείξει το Κοινοβούλιο προς αυτό το τομέα. Επίσης, η Αυστριακή Προεδρία θα ασχοληθεί με το θέμα των εμβολιασμών. Η πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία για την αντιμετώπιση των ασθενειών που μπορούν να αποτραπούν μέσω εμβολιασμών, σχεδιάζουμε να το συζητήσουμε τον Δεκέμβριο στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών. Επίσης, ιδιαίτερα φιλόδοξη στόχοι, συγγνώμη, υπάρχουν και σχετικά με την επικαιροποίηση του κανονισμού για τις γενικές αρχές της, του δικαίου για τα τρόφιμα. Εδώ έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε εντατικά τις ε, διαπραγματεύσεις έτσι ώστε το Νοέμβριο να έχουμε μια εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο, ε, οι διαπραγματεύσει του τριμερού διαλόγου που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια τη Βουλγαρική Προεδρία για τον κανονισμό για τα αλκοολούχα ποτά θα προσπαθήσουμε να τι ολοκληρώσουμε. Οι διαπραγματεύσει επίση για την οδηγία για, το, για τα πόσιμα ύδατα θα συνεχιστούν στην ομάδα εργασίας για το περιβάλλον. Η υψηλή ποιότητα του πόσιμου ε, νερού και, το, και, τα, και η ε, εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών βεβαίως πρέπει να είναι κάτι που θα μπορούμε να το εγγυηθούμε και στο μέλλον. Ε, βεβαίως υπάρχουν διάφορες δομές που ασχολούνται με τα, θέματα, με τα ή με τα υπόγεια ύδατα και βεβαίως θα τους δοθεί απαραίτητη προσοχή. Και ω προ αυτά τα θέματα η Αυστριακή Προεδρία θα συνεχίσει τι ε, διαπραγματεύσει. Επίση, η Αυστριακή Προεδρία θα αναλάβει την 8η διάσκεψη των ε, συμβαλωμένων μερών για, το, ε, για τη Συμφωνία Πλαίσιο για τον Καπνό. Σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατημέλη θα συνεργαστούν έτσι ώστε στη Γενέβη να μιλήσουμε με μία φωνή και να έχουμε μία συγκεκριμένη συμπεφωνημένη άποψη. Πέραν αυτού, στις 22 και στις 23 Νοεμβρίου θα κάνουμε μία ε, ε, τομεακή διάσκεψη για τα θέματα της ε, διατροφικής αλυσίδας και της προστιθέμενης αξίας. Ως προς αυτό, να ευχαριστήσω όχι μόνο την Βουλγαρική Προεδρία για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόθεση που έδωσε στο θέμα των τρανσλιπαρών οξέων. Ε, πραγματικά είναι σημαντικά, τα επιτέγματα αυτά που θα μας βοηθήσουν. Άλλο ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την Αυστριακή Προεδρία είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τους επόμενους μήνες θα γίνουν διάφορες συζητήσεις επί τη βάση διαφόρων τομεακών ε, γράφων στο Συμβούλιο. Τώρα, εγώ ως Υπουργό Κοινωνικών Θεμάτων και Θεμάτων Υγείας θεωρώ ότι η συμμετοχή του ε, προγράμματος δράσης για την υγεία θα, και η ένταξή του στην, ε, στο, στο μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus ε, τη βλέπω θετικά, γιατί αυτή η η συμπερίληψη μπορεί να αποτελέσει ε, θετική εξέλιξη. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε την ε, πτυχή της υγείας σε όλες τις πολιτικές και να μην την ξεχνούμε. Ε, θέματα που άπτονται της υγείας, πέραν του ε, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πλάς βρίσκονται και σε πολλά ε, τομεακά έγγραφα εντός του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για τον τομέα της υγείας υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ της παραδοσιακής υγείας, της βιωσιμότητας του δημόσιου προπολογισμού, καθώς επίσης και της οικονομικής πολιτικής ως προς την απασχόληση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Είμαι πεπισμένη ότι σε μια ενωμένη Ευρώπη μπορούμε μόνο με ε, μια ε, σταθερή ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία να προχωρήσουμε. Και ελπίζω ότι και εδώ μπορούμε να υπολογίζουμε στη δική σας υποστήριξη. Για το πρόγραμμα για την υγεία, για το περιβάλλον τώρα. Είναι μεγάλη χαρά που σε ό,τι αφορά την Προεδρία της Αυστριακής Προεδρίας ε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία συγκαταλέγονται στα πιο υψηλά του κόσμου και αυτό προφανώς είναι θετικό και είναι δύο οι λόγοι. Καταρχάς ε, για την προστασία της υγείας, της ε, ποιότητας της ζωής των πολιτών μας αλλά και για την προστασία της φύσης. Κατά δεύτερον, τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα εκ παραλλήλου δίνουν κίνητρα για την καινοτομία της πράσινης της απασχόλησης και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος της Τρόικας θα θέλαμε να συνεχίσουμε την επιτυχία και τις επιτυχίες εργασίες της Βουλγαρίας και να ανοίξουμε και νέους ε, φακέλους. Η προστασία του περιβάλλοντος και η κυκλική οικονομία κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας, όπως και στο παρελθόν άλλωστε, θα αποτελέσουν σημείο προτεραιότητας και πάνω απ' όλα είναι ο στόχος της εφαρμογής μιας βιώσιμη πολιτικής και της ατζέντα του 2030 στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας στην ε, ψήφιση το 2015 της συνθήκης του Παρισιού νομίζω ότι αποτελεί ένα πολιτικό ορόσημο στη φάση της εφαρμογής και υλοποίησης. Όλοι οι φορείς θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες στους επόμενους έξι μήνες. Η Αυστριακή Προεδρία λοιπόν θα ήθελα να συμμετέχει αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και τα κράτη-μέλη στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Η Αυστριακή Προεδρία λοιπόν τον Οκτώβριο θα υποβάλει τις προτάσεις μας τον Οκτώβριο του 2018 προκειμένου ε, στην COP24 ε, να τεθούν στο Κατοβίτς οι γραμμές, οι κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν στο Κατοβίτσι να πετύχουμε καλά αποτελέσματα για να έχουμε καταρχάς ε, υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας, κατά δεύτερον να είναι υλοποιήσιμα όλα αυτά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τρίτον οι διάφορες εθνικές ε, συνθήκες πλαίσιο να λεφθούν επαρκώς υπόψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την πρόθεση των κλιματικών στόχων σε διεθνές επίπεδο και η Αυστριακή Προεδρία στα πλαίσια της προετοιμασίας στο Κατροβίτς θα συνεχίσει τον στενό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερως μας απασχολεί στην Αυστριακή Προεδρέα η προώθηση των ε, υγιεινών συστημάτων μετακίνησης με περιορισμένη εκπομπή διοξιδίου άνθρακα. Και κοινός μας στόχο θα πρέπει να είναι η επένδυση και η κοινοτομία σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά τα οχήματα στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν και άρα τον επίσημο συνέδριο της 29ης Οκτωβρίου στην Αυστρία, στην πόλη μου Γκράτσα, θα τεθεί το θέμα αυτό ακριβώς ε, στο επίκεντρο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρότυπα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για τα γιοταχή και για τα υπόλοιπα οχήματα θα πρέπει να είναι υψηλή προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά την επίπεδο φιλοδοξία, υπάρχουν διαφορετικέ απόψει ε, στο Συμβούλιο. Ωστόσο, για ένα πράγμα συμφωνούμε. Θέλουμε στο θέμα αυτό να πετύχουμε μια συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε και αισιόδοξοι. στις 9 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο για το περιβάλλον θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε, θεωρούμε, μια απόφαση ό,τι αφορά το κλίμα. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε τρισμερής διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σκοπός μας είναι μέχρι τέλος του έτους να έχουμε πετύχει μια συμφωνία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το θέμα αυτό αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και όλος ιδιαίτερος ε, την κυρία Μαρέν την εισηγήτρια, για την δουλειά που έχει ήδη κάνει. Στην παρούσα φάση οι εκπομπές ε, βαρέων οχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ρυθμίζονται και αντιπροσωπεύουν παρόλα αυτά ένα τέταρτο του συνόλου των οδικών ε, εκπομπών και πρόκειται λοιπόν για μια δραματική αύξηση, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το 2030, μάλιστα, αν δεν δράσουμε όπως πρέπει. Θέλουμε λοιπόν να το ρυθμίσουμε το θέμα αυτό για να τηρηθούν και οι στόχοι που τέθησαν στη συνθήκη του Παρισιού. Θέλουμε να σημειωθεί πρόοδο ε, στο θέμα αυτό. Όσο πιο πολύ πρόοδο γίνεται και η Αυστριακή Προεδρία παρακολουθεί τι εργασίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Στα πλαίσια λοιπόν του προγραμματό τη Τροϊκά, η Αυστριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στην κυκλική οικονομία και κυρίω θα συνεχίσει το έργο σε ό,τι αφορά τα πλαστικά. Γιατί η Αυστρία εδώ και χρόνια σε ό,τι αφορά τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά δραστηριοποιείται και θέλει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική για το πλαστικό. Η Αυστριακή λοιπόν Προεδρία θέλει μεγαλύτερη δέσμευση κατά της ρήπανσης με πλαστικά και να δοθεί ακριβώς ε, προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Η πρόταση λοιπόν για μια οδηγία για τη μείωση των επιπτώσεων κάποιων πλαστικού στο περιβάλλον είναι για μας προτεραιότητα. Τα θέματα λοιπόν είναι τα εξή. Πώ μπορούμε η παραγωγή και η χρήση τέτοιων πλαστικών προϊόντων μια χρήση, τα οποία πετυχαίνονται μετά από μια χρήση δηλαδή, να περιοριστεί ε, με επιτυχία και πώ θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον και τι θάλασσές μα από τι αρνητικέ επιπτώσει των πλαστικών απορριμμάτων και πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τι πόρου μα και να προωθήσουμε τις οικολογικές προτεραιότητες και καινοτομίες. Οι συζητήσεις για τα πλαστικά μίας χρήσης έχουν ξεκινήσει ήδη στις προπαρασκευαστικές ομάδες του Συμβουλίου από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Φρεντερική η συγχύτρια, έχει ήδη κάνει πολύ καλή δουλειά είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φιλοδοξία μας δεν είναι μέχρι τέλος του έτους να έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο ό,τι αφορά το σημαντικό αυτό θέμα. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας ε, σε ό,τι αφορά κάποιες ε, οργανικές ε, επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες ονομάζονται POP, POPs. Αυτά τα χημικά λοιπόν, επειδή έχουν μεγάλη διαρκεία ζωή και είναι πάρα πολύ τοξικά, αποτελούν ένα ιδιαίτερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Η Αυστριακή Προεδρία λοιπόν καλωσορίζει ορίζει την πρόταση την οποία αναμέναμε πολύ καιρό για την ε, αναθεώρηση της σχετικού κανονισμού για τα POP, για τα χημικά αυτά. Η επεξεργασία λοιπόν, ε, η αναθεώρηση της ε, κανονισμού αυτό είναι απαραίτητη για να τηρηθούν οι συνθήκε και οι όροι τη συμφωνία τη Στοκχόλμη. Η Αυστριακή λοιπόν Προεδρία θέλει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχο μα στο θέμα αυτό είναι μέχρι τέλη του έτου να έχουμε πετύχει ε, συμφωνία σε πρώτη αναγνώση. Το δεύτερο ήμιση του 2018 θα περιλαμβάνει επίση πληθώρα δραστηριοτήτων για την προστασία των, της και της Προστασία τη φύση. Η Αυστριακή Προεδρία θα κάνει λοιπόν ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών σε διάφορε διεθνεί συναντήσει στον τομέα τη βιοπικιλότητα και τη προστασία τη φύση. Και τον Οκτώβριο θα έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ε, κατεύθυνση της μελλοντική παγκόσμιας πολιτικής για την βιοποικιλότητα μετά το 2020. Και έτσι λοιπόν δίνεται μια σημαντική έντολη για τις διαπραγματεύσει σε ό,τι αφορά το COP14, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τη βιολογική βιοποικιλότητα και για τη συμφωνία για τα δύο πρωτοκόλλα της συνθήκης. Η Αυστριακή Προεδρία καλωσορίσει επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδιαμόρφωση του πρόγραμματος LIFE μετά το 2020. Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιδοτήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εστιάζεται αποκλειστικά στο περιβάλλον, στο κλίμα και στην προστασία του, της φύσης. Το έτος 2020 θα σταματήσει λοιπόν η τρέχουσα πραγματική περίοδο. Οι εμπειρίε μας μας έχουν ε, διδάξει πολλά σε ό,τι αφορά και την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος LIFE. Θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο το μελλοντικό πρόγραμμα LIFE, γιατί στόχος μας είναι τους επόμενους έξι μήνες να σημειώσουμε όσο μεγαλύτερη πρόοδος γίνεται. Αυτό ασφαλώς εξαρτάται και από τις επραγματεύσεις για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ορίσει τα οικονομικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE. Η Αυστριακή Προεδρία θα ασχοληθεί και με άλλο ένα φάκελο, το οποίο ψηφίστηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την πρόταση την προσαρμογή των ε, διάφορων οδηγιών για το περιβάλλον. Αυτό θα περιορίσει λοιπόν το διοικητικό άχθος και έτσι θα προκύψει μια κατάσταση διπλού ωφέλους. Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε να σημειωθεί μεγάλη πρόοδος και στο θέμα αυτό τους επόμενους μήνες. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ένα πολύ αποτελετικό πρόγραμμα μπροστά μας. Ωστόσο είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι με στοχευμένη εργασία και με την καλό διάλογο και τη στενή συνεργασία θα πετύχουμε επίσης σημαντική πρόοδο για την ευημερία και την προστασία της ε, υγείας, του περιβάλλοντος και όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είναι χαρά μου να ακούσω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας και θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας ασφαλώς ε, όσο καλύτερα μπορώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Minister, for your presentation, ε, σας ευχαριστούμε πολύ, ε, κυρία Υπουργέ. Θίξατε πολλά θέματα, κάτι το οποίο δείχνει ότι γνωρίζετε πολύ καλά την ε, εργασία που μας απασχολεί και εμάς. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο με τους συντονιστές ή τους εκπροσώπους τους για δύο λεπτά τον καθένα. Ο Πίτερ Λίζε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα από τον τομέα της υγείας και ένα θέμα από τον τομέα της περιβάλλοντος. Καταρχάς, ε, στο βασικό ζήτημα του χαρτοβουλικής ύψας, ε, στο θέμα της υγείας. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι κάθε εβδομάδα στην Ευρώπη χάνουμε πολίτες, χάνουμε ανθρώπινες ζωές γιατί έχουμε βακτήρια τα οποία είναι ανθεκτικά στα Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε πολλά επίπεδα. Έχουμε την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα φάρμακα για τα ζώα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε και το θέμα των αντιβιωτικών για του ανθρώπου, Στην έκθεση τη κυρία Κάντνμπαχ πριν από κάποιες εβδομάδες αποφασίσαμε να ζητήσουμε νομοθετική πρόταση για την προώθηση νέων αντιβιωτικών. Γιατί ό,τι άλλο και να κάνουμε δεν επαρκεί θα συνεχίσουμε να χάνουμε ανθρώπινες ζωές αν δεν αναπτύξουμε νέα αντιβιωτικά. Και στην παρούσα φάση δεν υπάρχει οποιαδήποτε κίνητρο. Και άρα δεν προωθείται η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει διάφορα μέτρα, αλλά πολύ απλά δεν αρκούν όλα αυτά. Εσείς θα μπορούσατε να ταχθείτε λοιπόν προκειμένου να προκύψει νομοθεσία και θα προκαλούσατε μεγάλη έκπληξη γιατί το κόμμα σας θεωρείται ευρωσκεπτικιστικό και θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν ζητούσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομοθεσία. Είσαστε κατά. Κατά δεύτερον, για το μέλλον των περιβάλλοντο, μιλήσατε για τη συνθήκη του Παρισιού. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και στα κράτη-μέλη ασφαλώ. Και εκφράστηκε ένα υπουργό και είπε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε κατά 40% του στόχου του Παρισιού. Η κυρία Κόστινγκερ λοιπόν ε, γέννησε, α, συνέβαλε στην αύξηση των στόχων για τις ανανεώσιμες ενέργειες και υπάρχει λοιπόν αυτή η συζήτηση για να ξεπεραστεί το 40%. Δυστυχώ, τέτοια συζήτηση δεν γίνεται πουθενά αλλού στον κόσμο. Τι θα μπορούσε λοιπόν να κάνει η Αυστριακή Προεδρία προκειμένου να μην συζητήσει μόνο η Ευρώπη για μεγαλύτερες προσπάθειες, αλλά και άλλα κράτη να κάνουν πιο πολλές προσπάθειες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δεσμεύσεις στις οποίες ε, ανέλαβαν. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ, που παρευρίσκεστε εδώ η Αυστριακή Προεδρία αναλαμβάνει σε ε, ένα σημείο, μια στιγμή ζωτική σημασία κοντά στο τέλος της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου. Και όπως είπατε, έχουμε να κάνουμε με θέματα τα οποία θα θέλατε εσείς να ολοκληρώσετε από περιφαλοντικής πλευράς λοιπόν Δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό λόγω της περιπλοκότητας των θεμάτων. Αναφερθήκατε και στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα οχήματα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει. Θα ήθελα όμως να μιλήσω και για στήματα υγείας, γιατί έχετε και αυτό το χαρτοφυλάκιο Κατανοώ ότι η Προεδρία θέλει να συμπληρώσει τομείς που έχουν καλυφθεί από τη Βουλγαρική Προεδρία, αλλά θέλουμε να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι. Η Αυστριακή Προεδρία θα πρέπει να προβάλλει τις εύρωστες θέσεις μας ενώπιον του Συμβουλίου για να υπάρξει πλήρη συνεργασία και να αποφύγουμε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Εσείς προέχεστε από μια χώρα που εκφράζει ευρωσκεπτικισμό, αλλά θα ήθελα να είμαι σίγουρη για τη δέσμευσή σας. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις σας ως προς τα φαρμακευτικά σκευάσματα έτσι ώστε να μην υπάρχει έλλειψη κατανόησης στον τομέα της ε, υγείας και στα πλαίσια του ΠΟΗ σε σχέση με την περιεκτικότητα σε καπνό των προϊόντων. Γιατί η Αυστρία έπρεπε να απαγορεύσει τη χρήση τσιγάρου από τους ε, δημόσιους χώρους από το Μάιο, αλλά η κυβέρνησή σας ε, αθέτησε αυτή την υποχρέωση, κάτι το οποίο ορίστηκε από τους εμπειρογνώμονες ως μια μεγάλη καταστροφή στον τομέα της υγείας. Θα ήθελα να είμαι σίγουρη ότι υπό την προεδρία σας δεν θα ληφθούν τέτοιες ε, τέτοιες αποφάσεις υπέρ της βιομηχανίας καπνών και κατά των πολιτών. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ο κύριος Πιέκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, για αυτή την λεπτομεριακή παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ε, Αυστριακής Προεδρίας. Μιλάμε για πολλές προτεραιότητες, δέκα περίπου. Για μένα η πρώτη προτεραιότητα είναι ο εμβολιασμός ε, για λόγους προφύλαξης. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εμβολιασμού, κάτι το οποίο οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Και δυστυχώς τα κινήματα κατά του εμβολιασμού γνωρίζουν ανωδική πορεία. Σε σχέση με την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προτίθεται να κάνει η Αυστριακή Προεδρία σε σχέση με τα, τις ιατρικές μηχανές και τον ιατρικό εξοπλισμό. Τώρα, ως προς τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχουν αυτή την υποχρεωτική αξιολόγηση στα κράτη-μέλη ή θα υπάρχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση επί του θέματος. Αυτό είναι διφορούμενο διότι ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προσδοκίες των ασθενών και εδώ θα έχουμε να κάνουμε με μία πολύ μεγάλη επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών. Σε σχέση τώρα με τα φαρμακευτικά σκευάσματα και ιδιαίτερα τα αντιβιωτικά, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε πέρα αυτού του πλαισίου. Γιατί θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι συνήθεις, οι συνήθεις ασθένειες μπορούν να αντιμετωπιστούν συλλογικά. Ευχαριστούμε κύριε Πιέκα, κανένας από τους φιλελευθέρους. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητή Υπουργέ, θα ήθελα να σας θίξω ένα ζήτημα που είναι το 62 Δύο χρόνια πριν η Επιτροπή ε, έθιξε ένα θέμα ε, αναθεώρησης της χρήσης ε, του καδμίου και εδώ και 30 χρόνια το κάδμιο έχει απαγορευτεί σχεδόν από κάθε χρήση και γι' αυτό έχει μειωθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δυστυχώς όμως το καδμίο χρησιμοποιείται στα φυτοφάρμακα, κάτι το οποίο είναι επιζήμιο στην ανθρώπινη υγεία και φυσικά είναι και μεγάλος επιμολυντής. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη έκθεση σε καδμίο του γενικού πληθυσμού και θεωρώ ότι δυστυχώς δυστυχώς η χρήση και των φωσφορούχων ε, ουσιών σχετίζεται και με την υψηλή έκθεση σε κάδμιο. Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι πολίτες και ιδιαίτερα τα παιδιά εκτίθενται ιδιαίτερα. Νομίζω ότι μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση καδμίου στα λιπάσματα και αυτό αφορά και τις ε, ε, ουσίες φωσφόρου. Στη στιγμή όμως που δεν υπάρχουν ε, νομικές προαπαιτήσεις, κανένας δεν θα κάνει τις σωστές ε, επενδύσεις. Έχουμε μιλήσει για δραστική μείωση, την οποία υποστηρίζει η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως, δυστυχώς, ε, δυστυχώς έχουμε δεχτεί τα 60 μίλιγκραμμ μέχρι τώρα αλλά θα πρέπει να λάβουμε ότι έτσι θα δράσουμε επί του 8% των συνολικών προϊόντων της αγοράς, αλλά θα πρέπει να μειώσουμε περαιτέρω τη χρήση καδμίου στην γη, στην αγροτική γη. Ποια είναι η θέση σας, μπορούμε να φασιστούμε στην Αυστριακή Προεδρία για να αλλάξει η θέση του Συμβουλίου, έτσι ώστε να έχουμε ένα περιβάλλον που να είναι ελεύθερο από το κάδμιο. Ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Προεδρεύουσα, καταρχάς καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε που μας δίνετε την ε, δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί σας για τους στόχους της ε, Αυστριακής Προεδρίας. Για ένα θέμα που συχνά αναφέρω εγώ στην Επιτροπή εδώ, το είπε και ο συνάδελφος πιο πριν, το θέμα της μικροβιακής αντίστασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογεί ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον κάθε χρόνο 25.000 άνθρωποι ε, πεθαίνουν λόγω μικροβιακής αντίστασης των βακτηρίων. Ο, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας επίσης ε, ε, μιλά για εκατομμύρια θανάτους μέσα σε λίγες δεκαετίες στο μέλλον. αυτά είναι πραγματικά συγκλονιστικά στοιχεία σε σχέση με τα στοιχεία που έχουμε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποιεί ότι η αντίσταση αυτή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου στο μέλλον και επίσης ο Επίτροπος Ανδριουκάητης μίλησε σχετικά για το θέμα αυτό. Για ένα, ε, μίλησε για ένα τσουνάμι. Το θέμα αυτό, κυρίως στη Βόρειο ε, Αμερική και στην ε, Ευρώπη, είναι ένα θέμα που απασχολεί και μιλούμε για πραγματικά ανεύθυνη χρήση, κατάχρηση ίσως. Η προληπτική χρήση των αντιβιωτικών, ας για την υγεία των ζώων είναι ένα σύμπτωμα είναι σαφή συνέπεια της ε, κακής υγείας των ζώων και της ε, λοιπούς ε, πλημελούς προστασίας τους. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν η Αυστρική Προεδρία θα επιμείνει για καλύτερες πρακτικές και για καλύτερη προστασία των ζώων στο Συμβούλιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών για τα ζώα. Επίσης, η προστασία των ε, καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και η δημόσια υγεία θα μπορέσουν να, να προοδεύσουν επίσης. Γιατί νομίζω ότι αν αποφύγουμε την, τα προβλήματα που δημιουργούνται για τα ζώα θα μπορέσουμε να, έχουμε όλους, να τους έχουμε όλους κερδισμένους και για την πλευρά των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριος Πετιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και Ευχαριστώ την Υπουργό που παρευρίσκεται εδώ. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου για το γεγονός ότι θεωρείστε ευρωσκεπτικιστές ως προς τον εμβολιασμό αυτό. Μας το έχουν προσάψει και εμάς, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ελπίζω λοιπόν ε, αυτό να ισχύει και σε σας. Και θα ήθελα να σας υποβάλω μία ερώτηση γιατί μιλήσατε για ενισχυμένη συνεργασία για τους εμβολιασμούς. Εμείς συμμεριζόμαστε αυτή τη στρατηγική έτσι ώστε να φτάσουμε σε ε, μεγαλύτερη κάλυψη, γεωγραφική κάλυψη του εμβολιασμού. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ουσιαστικές συστάσεις και αυτή τη στιγμή 15 κράτη-μέλη δεν έχουν δεσμευτική προσέγγιση επί του θέματος των εμβαλιασμών. Όμως στην Ιταλία η προηγούμενη κυβέρνηση έλαβε μία, ένα δεσμευτικό μέτρο και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι προθέσεις αυτής της Προεδρίας. Θα ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να οθήσουμε τον πληθυσμό στον εμβολιασμό ή θα υπάρχει δεσμευτική προσέγγιση, γιατί αν υπάρχουν και οι δύο προσέγγισεις, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ενισχυμένη συνεργασία σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκοντίν. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Γκοντέν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ καταρχήν για το διορισμό σας και να σας πω ότι χαιρόμαστε εδώ που σας καλωσορίζουμε στα πλαίσια της Αυστριακής Προεδρίας. Έχω δύο ερωτήματα. Από το 2015 ο διαθεσμικός ε, διάλογος ε, για ε, την κλωνοποίηση των ζώων για γεωργικούς σκοπούς έχει απαγορευτεί για λόγους ηχνηλασιμότητας. Ε, Πρόκειται όμως για μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα πρέπει να ελέγξουμε ε, και το, τη χρήση αυτής της μεθόδου στις ε, εισαγωγές από τις τρίτες χώρες έτσι ώστε να έχουμε σαφή θέση. Αυτό θα είναι προτεραιότητα του Συμβουλίου. Δεύτερον, ως προς την πρόταση της Επιτροπής για τις ε, αξιολογήσεις των ε, τεχνολογιών υγείας, ιδιαίτερα τα άρθρα 8 και 22 που θέτουν θέμα επικουρικότητας και συρρυκνώνουν τις, ε, τη, θέση μας και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε επίπεδο Συμβουλίου ποιες είναι οι συστάσεις σας και οι θέσεις σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συμβουλίου. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και έτσι ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων. Τώρα δώσω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει στα ερωτήματα που ακούσαμε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ κύριε και κυρίες βουλευτές για τις ερωτήσεις σας και ελπίζω να μην ξεχάσω καμία. Κυρία Πρόεδρε, στην αρχή, στην εισαγωγή σας κάνετε και μία ερώτηση την οποία επιτρέψτε μου να απαντήσω στην παρούσα φάση. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Υγείας BMF+. Οι πραγματεύσεις για το BSF Plus θα είναι σίγουρα πολύ περίπλοκες γιατί περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα σε ό,τι αφορά συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε ό,τι αφορά το ξεχωριστό σκέλος για την υγεία. Οι συνέργειες και οι διαπαφές μεταξύ των προγραμμάτων υγείας και των άλλων προγραμμάτων θεωρώ ότι θα πρέπει να ειδωθούν σε ένα συνολικό συγκεκριμένο, γιατί μια ξεχωριστή αντιμετώπιση δεν θα ήταν χρήσιμη και στοχευμένη. Οι ειδικοί για θέματα υγείας φυσικά θα πρέπει να συμπεριλαμβανθούν και αυτοί. Για την ερώτηση του κυρίου Λίζα και του κυρίου Εκ, ο κύριος Λίζα, αν δεν κάνω λάθος, ε, ε, έφυγε σε ό,τι αφορά την αντιμικροβιακή αντοχή. Πρόκειται για μια παγκόσμια απειλή. Ω τέτοια αντιμετωπίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε για την αναθεώρηση της σχετικής ε, νομοθεσίας ε, σε ό,τι αφορά και τα αντιβιωτικά για τα ζώα, αλλά και κάποια κρίσιμα αντιβιωτικά για την ανθρώπινη κατανάλωση. Υποστηρίζουμε λοιπόν το, το σχέδιο δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου του 2017 για την αντιβιομικροβιακή ε, αντοχή και έγινε και το 2000, ε, θα προγραμματίσετε μάλλον και σε ένα σχετικό, μια σχετική ημερίδα για το θέμα αυτό. Μία άλλη ερώτηση του κυρίου Λύση, την οποία θα την απαντήσω παρά το γεγονό ότι έφυγε. Το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά πόσον ε, θα είχε νόημα να υπάρξει σχετική νομοθεσία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εξετάζουμε αυτό. Να ευχαριστήσουμε ωστόσο την κυρία Κάντενμπαχ και, Ευρωπαϊ... και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την σχετική έκθεση. Επίση, μία ερώτηση του κυρίου Νάλη και του κυρίου Παντιτσίνη και ελπίζω να μην κάνω λάθο στην προφορά των ονομάτων. Για το κατά πόσον το Συμβούλιο θα ακολουθήσει τι συστάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε, αντιλαμβανόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μας ενδιαφέρουν φυσικά τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τώρα τις προθέσεις του Συμβουλίου, ρώτησε η κυρία Τάλη, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων. Θέλω να είμαστε επικοδομητικοί σε ό,τι αφορά τις συστάσεις και κυρίως ό,τι αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για την επιτεύξη κοινών στόχων. Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμού, οι εμβολιασμοί είναι από τα πιο αποτελεσματικά προληπτικά μέσα τα οποία έχει στην της η... ο τομέας της υγείας. Υπάρχουν εθνικά μέσα για το θέμα αυτό για το θέμα της Αυστρίας. Ε. Η Αυστρία τηρεί και τις διεθνείς και τις εθνικές ε, προδιαγραφές σε ό,τι αφορά την υγεία. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ε, διεθνή εικόνα της Αυστρίας εδώ στη ΙΟΜΠΗ. Θέλουμε λοιπόν να μιλάμε με την αντίφωνη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Πιέκα έφτασε στο θέμα των εμβολιασμών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υποστηρίζουμε τις ε, ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά του εμβολιασμού. Και ο στόχος μας είναι κατά τη διάρκεια τη Προεδρίας να εγκρίνουμε το σχετικό κείμενο. Μια άλλη ερώτηση του κ. Πιέκα αφορούσε την πρόταση κανονισμού για το άρθρο 8. Προκειμένου η συζήτηση να συνεχιστεί και να συνεχιστεί μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο στις τεχνικές ομάδες του Συμβουλίου και να α, μπορέσουμε να κοιτάξουμε με επικοδομητικό τρόπο τα προβλήματα που έθεσαν τα κρατημέλη. θα κάνουμε ένα σωστό έλεγχο του σχεδίου νομοθεσίας. Δεν έχει νόημα λοιπόν στην παρούσα φάση να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Πρωτού η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ασχοληθεί με τους διάφορους ευρύτερους τομείς. Και οι διαπραγματεύσει ξεκινούν αύριο. Για την κυρία Άουκεν τώρα, για τα λοιπάσματα η Βουλγαρική Προεδρία στους τρομερείς διαολόγους ε, θεωρώ ότι σημείωσε μεγάλη πρόοδο και η Αυστριακή Προεδρία σκοπεύει να συνεχίσει έτσι δυναμικά και να συνεχίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Τίφεται και το θέμα του οριακών τιμών για το καδμίο και η ρήπανση αποτελεί, εξακολουθεί να αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την συνένεση και τη συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθεια σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πρώτων υλών, προκειμένου να κλείσουν τα θέματα αυτά σε πρώτη ανάγνωση. Για το θέμα της κλωνοποίησης, το έθεσε η κυρία Γκοντά. Η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κλωνοποίηση ζώων μας είναι γνωστή. Είμαστε ενήμεροι είναι γεγονό ότι οι διαπραγματεύσεις δεν σημείωσαν σημαντικό προ... σημαντική πρόοδο κατά το παρελθόν και ο λόγος για την έλλειψη αυτή επιτυχίας ε, των διαπραγματεύσεων είναι ότι η νομική βάση που επέλεξε η Κομισιόν και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου θεωρείται κατάλληλη και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή ε, η Αυστριακή Προεδρία δεν θα ακολουθήσει την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ωραία, περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων που θα καλύψει την υγεία και την ασφάλεια τροφίμων. Έχουν ε, εγγραφεί συνάδελφοι. Η κυρία Ζόμερ είναι η πρώτη ομιλήτρια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ. Ένα ερώτημα για τα τρόφιμα έχω να θέσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη τον Απρίλιο μας έκανε μια πρόταση για την νέα εκδοχή του βασικού κανονισμού επί του οποίου ε, περιμέναμε, για τον οποίο μάλλον περιμέναμε δύο, έξι χρόνια και είναι τώρα το τέλος της θητείας μας. Το ε, Συμβούλιο είναι υποπίεση και η Προεδρία του Συμβουλίου ε, πρέπει να τα κάνει όλα αρπακόλα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι. Η δική μου λοιπόν η ερώτηση είναι, η Αυστρία ως ευρωπαϊκή χώρα έχει κάποια θέση για την αναθεώρηση του βασικού κανονισμού για τα τρόφιμα και θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι η Αυστριακή Προεδρία θα τα καταφέρει να καταλήξει σε μια κοινή θέση του Συμβουλίου μέχρι το αργότερο του τα τέλη Νοεμβρίου για να μπορέσουμε τελικά στην πρώτη ανάγνωση να καταλήξουμε στη συμφωνία γιατί αλλιώς ο φάκελος ε, δεν θα προλάβει να περάσει πριν τις ε, ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ. Okay, thank Η κυρία Καμπεθόν. Ευχαριστώ πολύ την Υπουργό για την παρουσία της και χαίρομαι γιατί θα φτάσουμε σε ένα συμβασμό σε σχέση με την εξέλιξη και την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας. Γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και ανασφάλεια στο Συμβούλιο, αλλά και δυνατότητες που υπάρχουν για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στον τομέα υγείας και προϊόντων υγείας από τους πολίτες και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας στο Συμβούλιο. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει καθαρά ε, ρόλο διοικητικής υποστήριξης ενώ τα κράτη-μέλη να αναλάβουν ε, πλήρη δράση στον ε, τομέα αυτό μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας και για μια επαναξιολόγηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει προσαρμογή σε εθνικό επίπεδο αυτό πιστεύουμε ότι θα το επιτύχει το Συμβούλιο. Ως προς το δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα θεωρούμε ότι ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας δεν μας οδήγησε στο να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστούμε πολύ που θα προωθήσετε αυτό το θέμα κατά την εξάμεινη προεδρία σας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ζόμερ και πάλι. Η κυρία Ζόμερ. Α, ε, σας είχα πάλι στον κατάλογό μου γι' αυτό. Όσο το διερευνάτε αυτό, θα δώσω το λόγο σε κάποιον άλλον. Συγγνώμη. Ναι, ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Ένα ερώτημα έχω ακόμα Πάλι για τον κανονισμό για τα τρόφιμα. Τι άποψη έχετε κύριε Υπουργέ για τους ε, κανόνες ε, για την καλύτερη ε, διακυβέρνηση. Ακόμη δεν έχουμε κάνει αξιολόγηση αντικτύπου και πρέπει να δούμε στο κενό και να επεξεργαστούμε τον κανονισμό αυτό και μιλούμε και για τον κανονισμό για την ενημέρωση των, των καταναλωτών. Ήδη υπάρχει από το 2011, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς και εν τω μεταξύ ερμηνεύεται με τα κράτη-μέλη ε, με τέτοιο τρόπο, ώστε ε, μπορούν τα κράτη-μέλη να φτιάξουν το δικό του σύστημα επισήμανσης, ε, το οποίο σιωπηρά το επιτρέπει η Κομισιόν. Αλλά αυτό είναι και επιθετικό και αρνητικό προς την ιστορική αγορά. Οπότε η Αυστριακή Προεδρία έχει υπόψη της να ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να το πράξετε. Ευχαριστώ. Uh, Η κυρία Κάντεμπαχ, καλώ ήρθατε κυρία Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Τα εισαγωγικά σα σχόλια είπατε ότι θέλετε να συμβάλλετε στην Ευρώπη, θέλετε να ενισχύσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλετε να αποκαταστήσετε την ε, εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες και εδώ στον οίκο μα και στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Υπάρχει ο η συγκεκριμένη νομοθεσία από την Αυστρία, η οποία δεν νομίζω ότι θα ταιριάξει την, με το όραμα που έχετε. Ε, και επίσης δεν νομίζω ότι θα είναι καλή η εκπροσώπηση στην διάσκεψη για τον, ε, ε, για τον καπνό. Έχουμε έναν, μια, δήλωση στον τύπο από τον Χάραλτ Βιλίμσκι, ο οποίο είναι κομμάτι της κυβέρνηση και λέει ότι εγώ καταψήφισα της, την διάσκεψη του για το κλίμα και η κυρία Κιώστιγκερ, η οποία επίσης είναι μέλος κυβέρνησης, λέει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση η ανευθυνότητα. Τι θέλετε ακριβώς, πώς θέλετε ακριβώς να έχετε ε, θέση ενιαία απέναντι ε, στα 27 κρατημέλη όταν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενιαία θέση εντός της δικής σας κυβέρνησης. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Και μάλιστα στην Επιτροπή σήμερα ε, δεν νομίζω ότι έχετε και πολλούς φίλους όταν μας λέτε ότι δεν θέλετε να έχετε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα υγείας. Η Επιτροπή μας γι' αυτό πολεμάει, γι' αυτό αγωνίζεται. Το είπε και η Πρόεδρος στην αρχή. Εμεί θέλουμε μια ενωμένη, ενισχυμένη Ευρώπη και για τον τομέα της υγείας. Αλλά ακριβώς αυτό είπαμε ότι δεν θέλουμε, γι' αυτό είπαμε ότι δεν θέλουμε το τομέα τη υγεία να μπει στον ε, γενικό προπολογισμό. Όταν κάνετε λοιπόν, είναι τελείω αντίθετο με αυτά που λέτε ότι θέλετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Ξέρετε, συνάδελφοι, τον κανόνα για, τους, ε, για το χρόνο ομιλία. Δεν, όσο παθιασμένη και αν είναι η παρέμβασή σας, δεν θα πάρετε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Η κυρία Όκεν. Thank you very much. And question proposal. Ε, ήθελα να μιλήσουμε ε, για τη διαφάνεια που υπάρχει στην αλυσίδα τροφίμων. Τώρα έχουμε μία με, μεγάλη βελτίωση στον τομέα της ε, διαφάνειας, αλλά όταν δούμε την ουσία βλέπουμε ότι αλλάζοντας το κατάλογο των ε, στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα. Τώρα έχουμε περισσότερους τομείς εμπιστευτικού χαρακτήρα. Μιλάμε για τα εμπορικά προϊόντα. Η Επιτροπή δεν αναφέρεται ούτε καν ε, στο θέμα του συμφέροντος, του δημοσίου συμφέροντος. Και αυτό αφορά και ε, μέρος μάλλον εντάσσεται στη Συμφωνία του Άρχους. Θα πρέπει να σταματήσουμε κάτι τέτοιο γιατί υπάρχει συρρήκνωση διαφάνειας. Έχουμε λιγότερη διαφάνεια και ξέρω, επειδή βρίσκομαι χρόνια στην πολιτική, γιατί ε, ξέρω, ακριβώς επειδή βρίσκομαι χρόνια στην πολιτική, ότι η διαφάνεια δεν είναι ένα ενιαίο θέμα. Υπάρχει πολύ λιγότερη διαφάνεια τώρα και ελπίζω βλέποντας ε, τον ε, κατάλογο να λάβετε υπόψη το συμφέρον του κοινού, το περιβάλλον και τα τρόφιμα και να μην δώσει το προβάδισμα στις βιομηχανίες τροφίμων. Ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ, είμαι υπεύθυνο ε, του προγράμματος υγείας και παρόλο που είναι ξεχωριστό από το ESF Plus είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ως προς την έρευνα έχει αυξηθεί κατά ένα εκατομμύριο θα προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε τις αποστολές, το ρόλο των αποστολών και το ρόλο του Κοινοβουλίου και των ε, κρατών μελών. Επίσης, ως προς την υπατήτηδα, ξέρω ότι θα υπάρξει μία εποπτεία και τα στοιχεία αυτής της επόπτευσης θα αποσταλούν τον Νοέμβριο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση εάν θέλουμε να εξαλειφθούν η υπατήτηδα στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκούτελαντ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Διάβασα το πρόγραμμα της Προεδρίας και άκουσα την ε, παρουσίασή σας με μεγάλη προσοχή. Χαίρομαι γιατί θέλετε να συνεχίσετε τη δραστηριότητα αυτή για τα POPs. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για την υγεία και για το περιβάλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μεγάλη επίπτωση αυτών των ε, διαταρακτών και υπάρχουν έχουν ε, συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια σε σχέση με τις ε, βιοκτόνες ουσίες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες ουσίες ε, πέρα από τα πλαστικά. Η Επιτροπή θέλει να υπάρξει ένα οριζόντιο ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε όλες τις κατηγορίες. Χρειαζόμαστε μια σαφή στρατηγική σε σχέση με ε, αυτούς τους ε, ορμονικούς διαταράκτες. Και δεν εδόθη απάντηση από το Διευθυντήριο των Επιτρόπων ο αντιπρόεδρος Κατάινεν που έχει την ε, αρμοδιότητα επί του θέματος δεν μας έχει απαντήσει. Τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει. Ωραία, έτσι τελειώνει και ο δεύτερος γύρος. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς για την ερώτηση της κυρίας Ζόμερ για το Γενικό Νόμο για τα Τρόφιμα. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για να υπάρχει διαφάνεια και αξιοπιστία σε ό,τι αφορά των αποτελεσματών των ερευνών. Και θέλουμε να προχωρήσουμε το των δυνατών τις εργασίες στο Συμβουλίο, προκειμένου να έχουμε σχετική εντολή και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε μέχρι το τέλη της Προεδρίας μας να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα θέλουμε να κάνουμε αυτά μέχρι τον Νοέμβριο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα τη κυρία ε, Σόμερ, σε ό,τι αφορά την προπαρασκευαστική επιτροπή του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά αυτό το γενικό νόμο για το τρόφιμα, ξεκίνησε τι εργασίε του και κάνει και μία μελέτη αντικτύπου η οποία θα ληφθεί υπόψη και στους κόλπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τη σήμανση, την εθνική σήμανση ανά χώρα δηλαδή. Και σε ό,τι αφορά την αναρμόνιση. Ε, Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει σημαντικό ε, βήμα. Η κυρία Καμπαστόν Ρουίς για το HTA. Ενίσχυση λοιπόν τη συνεργασία σε ό,τι αφορά το HDA, την αξιολόγηση τέτοιων ε, μηχανημάτων υγεία είναι προ το συμφέρον και τη υγεία των ασθενών και του περιορισμού του κόστους. Θα συζητηθεί αυτό και στις 22... Συζητήθηκε μάλλον αυτό και στις 22 Ιουνίου στο Σχετικό Συμβούλιο Υγείας. Υπάρχει λοιπόν αντατική και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με στόχο το συντομότερα δυνατόν να πετύχουμε όσο μεγαλύτερη πρόοδο γίνεται. Όπως για παράδειγμα μια τομεακή κατεύθυνση. Το θέμα της κυρίας Κάρνμπαχ το θέμα του καπνίσματος. Να με αξιολογήσετε βάσει των πραξεών μου, σας παρακαλώ, για την κυρία Άουκεν. Ξέρουμε ότι χρειάζεται το συντομότερο δυνατόν μία απάντηση για τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Πολίτη για την διαφάνεια και την αξιοπιστία του, των ερευνών σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και θα μπορέσουμε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να προωθηθούν οι εργασίες αυτές όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Συμβούλιο. Το θέμα των συστάσεων για τον εμβολιασμό αποτελεί θέμα προτεραιότητας και σίγουρα θα μας απασχολήσει. Για την κυρία Κούτελαντ να πω ότι η Αυστριακή Προεδρία χαίρεται που θα ξεκινήσει όσον ούπο τι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ε, τροποποίηση των κανονισμών για τις ε, τοξικές αυτές ουσίες και προκειμένου να προσαρμοστούν οι υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στη συνθήκη της Στοκόλμης και σκοπεύουμε μέχρι τέλους του έτους να πετύχουμε αν γίνεται συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και περιμένουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά και ένα από τα προσαρτήματα της συνθήκης της Στοκχόλμης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και τώρα κάποιες ερωτήσεις έχουμε για το περιβάλλον και το κλίμα. Ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για τη διαθεσιμότητα μπροστά σας ε, για να απαντήσετε και θέματα που δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας. Ευχαριστούμε που αντικαταστήσατε την Ελίζαμπετ Κέστιγκερ. Είπατε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Αυστριακής ε, Προεδρίας είναι και η οδηγία περί υδάτων. Ξέρετε ότι πρόκειται για ακριβοθόρητο ε, αγαθό, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες και περιοχές του νότου της Ευρώπης. Μέσα στα πλαίσια της ρυθμιστικής αναθεώρησης για την ποιότητα των υδάτων υπάρχουν και στοιχεία πολύ ευαίσθητα. Ο ΠΟΗ μιλάει για 2,4 μιλιγκράμμ ανά ε, λίτρο. Αλλά για να είναι το νερό ε, πόσιμο θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσο υπάρχουν ε, στοιχεία ηλίως τα οποία βρίσκονται κάτω από αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο θα συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε την ε, προληπτική αρχή για να έχουμε νερό το οποίο να είναι πραγματικά διαθέσιμο, πόσιμο και καθαρό. Η κυρία Γκούτελαντ. Ευχαριστώ. Και εγώ με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να μιλήσω για την ε, βιοοικονομία. Τι ακριβώς ε, προτίθεται να κάνει η Αυστριακή Προεδρία. Η βιοοικονομία έχει μεγάλη σημασία για τα δάση μας. Και εδώ υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ Αυστρίας και δικής μου χώρας. Τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τις πλαστικές και χημικές ε, ύλες και ουσίες. Τι μπορούμε να κάνουμε με την κυκλική οικονομία. Μπορούμε να μιλάμε για πολιτική κλίματος, υπέρ του κλίματος, χάρη στα δάση μας, που είναι οι μεγάλοι μας πνεύμονες. Πώς θα προωθήσετε αυτήν την εργασία και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας σε σχέση με την εποπτεία των δασών. Επίσης και κάτι, και κάτι άλλο το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα. Η χρήση των λιπασμάτων. Η βιώσιμη χρήση των λιπασμάτων. Μιλήσατε για μία εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει μεγάλη σημασία και για την ΚΑΠ αλλά και για τα δάση. Ποια είναι η θέση της Αυστρίας για να υπάρξει σωστή εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Δεμεσμάκερ. Σας ευχαριστώ και καλώς ορίσατε κυρία Υπουργέ. Να σας ε, Ευχηθώ και κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω. Η μία για την βιοπικιλότητα και μία για την κυκλική οικονομία. Βιοπικιλότητα. Χαίρομαι που προετοιμάζεστε για μια πολιτική για την βιοπικιλότητα μετά το 2020 και που υποστηρίζετε τις ε, πολιτικές αυτές. Ελπίζω όμως η φιλοδοξία να είναι λίγο πιο υψηλή από αυτές που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, σε ό,τι αφορά το μελλοντικό πρόγραμμα LIFE η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λοιπόν την φιλοδοξία να σταματήσει να ανακόψει την απώλεια βιοπικιλότητα, γιατί περνάει κρίση βιοπικιλότητα. Αν θέλουμε λοιπόν να εκπληρώσουμε αυτή την φιλοδοξία, χρειαζόμαστε πολύ απλά και τα εργαλεία και έναν αντίστοιχο προπολογισμό. Και πολύ φοβάμαι ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι αφορά το θέμα αυτό υστερεί. Υστερεί σημαντικά. Ελπίζω αυτό να εννοήσατε όταν είπατε εισαγωγικά ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς απο... ένα πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα live. Ελπίζω να είμαστε σύμμαχοι, να είστε σύμμαχο ε, δικό μα σε ό,τι αφορά την αύξηση τη χρηματοδότησης χρηματοδότηση. Κυκλική οικονομία. Η, η έκθεσή μου για τα πλαστικά σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκε εδώ στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα πλαστικά μια χρήση. Ε, Χαίρομαι που το θίξατε το θέμα αυτό, αλλά είπατε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει πιο πολύ πλαστικό μιας χρήσης στην κυκλοφορία. Πιστεύετε ότι είναι λογικό να χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και μπορούν να αντέξουν για μία ολόκληρη ζωή για πάντα. Θεωρώ ότι θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε πιο λίγα μικροπλαστικά, πιο λίγα πλαστικά και ελπίζω πραγματικά και εκεί να είστε σύμμαχο δικό μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Παλούτσι, τελευταίος. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Τους επόμενους μήνες θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε το θέμα και ε, εγώ είμαι εισηγητής και όδηση εισηγητής για τη χρήση των ε, πλαστικών μίας χρήσης. Θα πρέπει και το Συμβούλιο να αναλάβει ευθύνες καθώς και η Προεδρία. Εσείς αναφερθήκατε στο θέμα αυτό προτεραιότητας έτσι ώστε να φτάσουμε σε ουσιώδη, σε ουσιώδη πρόοδο μέχρι το τέλος του έτους. Θεωρείτε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία ε, κοινή θέση με το Συμβούλιο για τη χρήση πλαστικών μίας ε, χρήσης. Μπορούμε να αρχίσουμε τους τριμερείς το Νοέμβριο. Ποιες, ποια είναι τα βασικά θετικά στοιχεία που υπάρχουν και Πού θεωρείτε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να υποβάλει κάποιο ερώτημα ή να κλείσω τον κατάλογο. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Α, η κυρία Κάντενμπαχ, αλλά για ένα λεπτό και επιμένω σε αυτό. Ανακοινώσατε ότι θα μας υποστηρίξετε στο θέμα της επισήμανσης ε, της νέας ε, τεχνολογίας για τη γενετική. Οπότε πώς ακριβώς ε, θα συμβάλλει στους επόμενους έξι μήνες η Αυστριακή Προεδρία για το θέμα αυτό της επισήμανσης της τεχνολογίας για τα γενετικά θέματα. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι. Κυρία Υπουργέ, σας ακούμε. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε για το ερώτημα για την οδηγία για το πόσιμο είδωρ. Ευχαριστώ καταρχάς για το ερώτημα. Το θεωρώ και εγώ πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η Αυστριακή Προεδρία θα ε, προχωρήσει τις εργασίες στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό και θα βασιστούμε βεβαίως και στην δουλειά των προηγούμενων μηνών και στις ε, δηλώσεις ε, του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου. Είναι σκηνό αυτό το, αυτή η ανησυχία ότι πρέπει να είναι καθαρό το νερό και υψηλή ποιότητα και βεβαίως πρέπει να δούμε τι γίνεται με την προστασία από επιμολυντικές ουσίες. Για την ε, ερώτηση Γκούτελαντ, για την ε, βιοοικονομία. Ε, εδώ υπάρχει πολλή δουλειά που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κίνητρα για διάφορους τομείς, για τα δάση και τη δασοκομεία θα σας την, θα παραπέμψω την απάντηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η Επιτροπή εδώ υπεύθυνη. Για το ερώτημα για το ΙΝΚΟΠ 14 Εκεί θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις για το θέμα της βιοπικιλότητα και της προστασία της φύσης. Η Αυστριακή Προεδρία θα ε, μπλακεί ενεργά και βεβαίω θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της σε αυτή την ε, διεθνή εκδήλωση. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να δούμε τα θέματα της βιοπικιλότητας, και βεβαίως θα δούμε την, ε, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα για την υπογραφή ε, των, ε, με, τα με τα συμβαλόμενα μέρη. Ελπίζουμε τον Οκτώβριο να έχουμε συμπεράσματα Συμβουλίου έτσι ώστε να έχουμε μια στεναρή διαπραγματευτική θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να είμαστε έτοιμοι για την στρατηγική για το πλαίσιο βιοπικιλότητας μετά το 2020. Άλλο ένα ερώτημα για το πρόγραμμα LIFE. Το Συμβούλιο ασχολείται αυτή τη στιγμή με την τεχνική συζήτηση της, ε, ε, ε, της πρώτης κομισιόν για το Live μετά το 2020. Επί τη βάση λοιπόν των αποτελεσμάτων από την διάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος προγράμματος LIFE θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για την μεθεπόμενη περίοδο έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική χρηματοδότηση για το κλίμα, την, τα βιώσιμα προγράμματα για την ενέργεια και η Αυστριακή Προεδρία το επόμενο εξάμεινο θα, κάνει, θα βάλει τα δυνατά της για να καταλήξουμε την, στην ολοκλήρωση του κανονισμού. Θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο βεβαίω θα, έχει την, θα έχει σημαντική επιρροή στο πώ θα δομηθεί το επόμενο πρόγραμμα LIFE. Άλλο ένα ερώτημα για το θέμα των πλαστικών μια χρήση. Η Αυστρική Προεδρία βεβαίω χαιρετίζει την τελευταία πρόταση για την οδηγία για τη μείωση τη χρήση σε συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων και την επιρροή του στο, στο περιβάλλον. Ε, και είναι πραγματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα έτσι ώστε να, μειωθεί και να μειωθούν τα απόβλητα πλαστικών και βεβαίως υπάρχουν κεντρικές πρωτοβουλίες ε, για την κυκλική οικονομία σχετικά. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν ως ε, μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας ε, να έχουμε γρήγορα βήματα προς τα εμπρός για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και είμαστε έτοιμοι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσουμε και εναλλακτικέ λύσεις έτσι ώστε στο τέλος, μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κατηγορίες των πλαστικών προϊόντων και τις διάφορες απαγορεύσεις, το Συμβούλιο και η Κομισιόν μελετούν την πρόταση και βεβαίως ε, θα δούμε τι θα γίνει και με την αξιολόγηση αντικτύπου. Για την, πάλι για το ερώτημα το, για τα πλαστικά. Όπως είπα θέλουμε γρήγορα να δουλέψουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ευρεία υποστήριξη. Για την κυρία Κάντενμπαχ. Το Συμβούλιο το, ε, και Αλίας τον ε, Ιούλιο του 2015 ε, έκανε μια συζήτηση. Από τότε δυστυχώς δεν έχουν ε, επανέλθει στο θέμα αυτό και από τότε ισχύουν τα αποτελέσματα. Η πλειοψηφία των κρατών μελών βεβαίως έχει προ, προσπαθεί να καταλήξει σε μια πρόταση. Το Κοινοβούλιο έχει απορρίψει την πρόταση που υπήρχε. Μέσω λοιπόν αυτής της πρότασης που έχουμε δεν έχουμε ασφάλεια δικαίου για, την, ε, για τους οργανισμού. τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου διατηρεί τη θέση που είχε και, η Ευρωπαϊκή, ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα κράτη-μέλη έχουν απορρίψει την πρόταση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει νέα πρόταση. Οπότε υποθέτουμε ότι οι διαπραγματεύσει για το θέμα αυτό δεν θα έχουν επιτυχή ε, κατάληξη. Οπότε δεν θα συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Well, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κύριε Υπουργέ, πολλά θέματα, πολλή εργασία μπροστά μας. Η Επιτροπή μας επίσης είναι αποφασισμένη να προωθεί στα ζητήματα αυτά χρόνο με το χρόνο. Ελπίζω να μας υποστηρίξετε σε θέματα υγείας έτσι ώστε να υπάρχει μια διαφορετική εγγραφή για το πρόγραμμα αυτό για να έχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα το ίδιο το πακέτο. Καταλαβαίνω ότι εσείς ασχολείστε και με τις κοινωνικές υποθέσεις και γι' αυτό θα είναι μεγάλη πρόκληση για μας να σας πείσουμε για θέματα υγείας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας, ε, ευχαριστού... και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία με την Προεδρία σας. Uh, we have a joint meeting with Στι 4.30 συνάδελφοι έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΤΕΒΕ για του ε, βιώσιμους στόχου.